Συνάδελφοι, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ελπίζω όλοι να περάσατε όμορφα το καλοκαίρι σας. Δύο σημαντικά θέματα έχουμε στη μερίσια διάταξη. Έχετε το σχέδιο μερίσια διάταξη μπροστά σα. Ε, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ωραία. Ε, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα πρακτικά της ε, συνεδρίασης ε, της 12ης και 13ης Ιουλίου. Να σας ρωτήσω αν μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Ωραία. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Προχωρώ στο θέμα 3, που είναι ο προϋπολογισμός για το 2011. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και κατόπιν θα ψηφίσουμε μετά την εξέταση των τροπολογιών. Δίνω λοιπόν το λόγο στον ε, εισηγητή μας για τον προϋπολογισμό, Ντομινίκ Ρικέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα αγόμεθα στο να συζητήσουμε και ψηφίσουμε ταυτόχρονα για λόγους ε, διαδικαστικής οικονομίας αυτή την έκθεση επί του προϋπολογισμού του 2011 που αφορά τις μεταφορές του τουλεχθέντος το Συμβούλιο απεφάνθη σε πρώτη ανάγνωση και επιβεβαίωσε μαζί με το Κορεπέρ ήδη από μήνος Ιουλίου. Η Επιτροπή του υπολογισμού θα αποφανθεί επί του συνόλου των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί μεταξύ των οποίων και αυτών τη επιτροπή μας την 28η, 29η και 30η προσεχού Σεπτεμβρίου. προθεσμία έχει τεθεί μέχρι 8 Σεπτεμβρίου για τους μεμονωμένους και τις πολιτικές ομάδες και ε, για την Ολομέλη θα περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Εκεί θα υπάρξει μία μόνο ανάγνωση, όπω γνωρίζετε. Οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου, όπω έχουν προσδιοριστεί από την ομάδα αξιολόγηση για το Τρίλογο, έχουν ήδη από 7 Ιουνίου ε, εγκριθεί με μια σειρά από σημαντικέ επικεφαλίδε, ειδικά η ΑΑ που μα ενδιαφέρει προκειμένου για το πολιετέ οικονομικό πρόγραμμα για τι μεταφορέ και τον τουρισμό. Οι συγκεκριμένε επιπτώσει για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι τη τάξη των 60 εκατομμυρίων ευρώ για την σταθεροποίηση, η χρηματοδότηση τη στρατηγική, το πρόγραμμα για την νεότητα, η θέση σε ε, ε, λειτουργία του εξωτερικού δικτύου, η αναθεώρηση του ΕΜΦΕΦ και των προβλημάτων που έχουν επιπτώσει στον προπολογισμό επίση. Τροπολογίες που αφορούν τη μεταφορά και τον τουρισμό ε, σε επίπεδο σπαντά ε, προτεραιότητες που μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο της αξιολόγηση και προαναγγέλλονται δυσχερείς. Οι προτάσεις ε, για τον προπολογισμό μεταφορών και τουρισμού συνήθανται στην πρόταση προπολογισμού ρεαλιστικού όσον αφορά την ε, προπολογιστική πειθαρχία. Και αυτή είναι η δική μα δουλειά. Εάν πρέπει να πούμε ότι η προηγούμενη μας έκθεση ε, έγινε καλά αποδεκτή και από την Επιτροπή του Προεπολογισμού και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό συνέβη γιατί η γενικότερη ενότητά μας η ΑΑ έχει περιοριστεί ως προς ε, τις πιστώσεις πληρωμών και τις εγκρίσεις προγράμματος ε, κατά 10% περίπου, ουσιαστικές περικοπές για τη μεταφορά, επιτύχαμε αύξηση παρά τα αυτά της τάξης του 9%. Αν μη τι άλλο, με τον τρόπο αυτό έχουμε κάποιο προνόμιο, έχουμε ευνοηθεί σε ένα γενικότερα δυσχερές συγκυριακό πλαίσιο. Όσον αφορά το κείμενο των προτάσεων, η έκθεση προσπαθεί να προτείνει συγκεκριμένες και όσο πιο συνεκτικές, συνοπτικές ε, ιδέες. Πρέπει να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται σε αυτό. Αποφύγαμε να προτείνουμε πράγματα ε, ε, ιδιαίτερα αναλυτικά, απλά στοχεύσαμε τα σημεία εκείνα που για μας κρίθηκαν πιο ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τα προεκτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ε, περιοριστήκαμε στα όσα είχαν εγκριθεί από τους συντονιστέ τη Επιτροπής μας και την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει δυνατότητα της τάξης των 120 εκατομμυρίων ευρώ έως και 50 ε, εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχω για τα προπαραγγελματικά και τις ενέργειες όπως επίσης και τα 300 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κατατεθεί από διάφορες επιτροπές Θεωρώ λοιπόν ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτά που οι συντονιστέ τη Επιτροπή μα είχαν προσδιορίσει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι διάφορε ομάδε μετά και από τι συζητήσει. Για τον λόγο αυτό, οι προτάσει παραμένουν στοχευμένε στι ε, ε, προτάσει δράσεων που είχαμε αρχικά αποφασίσει. Συνολικά, μιλάμε για 3 εκατομμύρια 800.000 για τα αγροπαρασκευαστικά, κάτι που αντιπροσωπεύει αναλογία της τάξης των 6% προκειμένου για ε, τις, το σύνολο των δράσεων των διαφορών προγραμμάτων. Όσον αφορά το σχέδιο υπερβολισμού των μεταφορών, ε, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στου οργανισμού, μια και αυτή είναι και η ισχυρή ε, ομάδα μα, ε, το ισχυρό κομμάτι της ομάδας μας. Το ίδιο σημαίνει και για τι διάφορε οργανώσει. Εδώ έχουμε μια χρόνια έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Οι τροπολογίε λοιπόν, που έχουμε προτείνει καταρχήν προσπαθούν να ισοσταθμίσουν τον προπολογισμό που προτείνει το Συμβούλιο να εξηγήσω ότι όλοι οι οργανισμοί από κοινού συζήτησαν το ζήτημα με μας ε, σε μια προσπάθεια εξέβραση μιας ισορροπίας μεταξύ των ε, τιμάτων, των αναγκών και των τελικών πραγματικών δυνατοτήτων που έχουμε για χρηματοδοτήσεις. Οι τροπολογίες που έχουμε προτείνει λοιπόν ως προς αυτό έτυχαν ε, τις εγκρίσεως εντός εισαγωγικών των οργανισμών έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας επαρκής προϋπολογισμός ε, όσον αφορά ε, διάφορα κονδύλια ε, και κάποιες προτάσεις που δεν μπορούν να αποδεχτούμε από πλευρά Συμβουλίου όσον αφορά τις ε, λειτουργικές δαπάνες άλλες πάλι μπορούν να προταθούν κυρίως σε επίπεδο διοικητικών δαπανών ε, οι περικοπές που αφορούν την ασφάλεια των μεταφορών το τα δικαιώματα των ε, επιβατών κτλ μπορούν να γίνουν αποδεκτές όσον αφορά την πρόταση για μια αρκετά ολοκληρωμένη ή κάποτε ακόμα και μερικώς ε, εξασφαλιζόμενη κατάσταση του προπολογισμού. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι εάν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, λίγο πολύ η, η θέση θα είναι αρκετά ικανοποιητική ε, στους κόλπους της Επιτροπής ε, του Προπολογισμού και στην ε, Κομισιόν. Το Συμβούλιο έδειξε μια κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τον ε, προπολογισμό των ε, μεταφορών, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα, μια και είναι γενικότερο το κείμενο, γενικά το δύσκολο το κείμενο, καλά έχουμε πάει. Αυτά εν είδη προημίου. ευχαριστώ πολύ. Ε. Ευχαριστώ πολύ, και Να ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτα έχουμε τον κύριο Βεράσκη για την ομάδα των σοσιαλιστών. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ο, ο εισηγητής μας, Ντομινίκ έχει κάνει πολλή δουλειά προσπαθώντας να βρει λύσεις που θα ωφελήσουν τον προϋπολογισμό της Επιτροπής μας. Όλα αυτά νομίζω μπορούμε να τα δεχτούμε. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ο προϋπολογισμός μας όλο και περισσότερο αρχίζει να μοιάζει με τους προϋπολογισμούς, με τους σχετικούς εθνικούς προϋπολογισμούς. Έχουμε αύξηση των σταθερών δαπανών για ε, νέες πρωτοβουλίες. Ενώ υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ε, που έχουν όλο και λιγότερη σημασία στο προπολογισμό, ενώ όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις ε, ή ε, τα θεσμικά όργανα αυξάνονται οι σχετικές δαπάνες και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ο κύριος Ρικέ έχει προγραμματίσει μεγάλο αριθμό συναντήσεων είχε προγραμματίσει μεγάλο αριθμό συναντήσεων για να διαπραγματευτεί και έδωσε επίσης χώρο διαπραγματευση στι πολιτικέ ομάδε για να καταλήξουμε ε, στην τελική μορφή του προπολογισμού όπου κάτι τέτοιο μπορούσε να ε, αιτιολογηθεί. Οι προτεραιότητε που περίμενε η πολιτική μου ομάδα πράγματι έχουν τεθεί. Καταρχήν λοιπόν το, ο προπολογισμό αυτός μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε βήμα-βήμα για να πετύχουμε ε, τον στόχο της ε, ολοκλήρωσης ε, και για να μπορέσουμε να ζητούμε όλο και περισσότερη δουλειά από τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούμε. Έχουμε καταλήξει σε αριθμό συμβιβασμών. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εύκολοι. Ιδιαίτερα ο πρώτος συμβιβασμός δεν ήταν εύκολος, εύκολο να επιτευχθεί και θέλαμε το διπλάσιο ή τριπλάσιο ποσό για την εφαρμογή του σχεδίου. Το συγκεκριμένο ποσό όμως ε, που αναφέρεται τελικά είναι αυτό που είναι σκόπιμο για την εφαρμογή του έργου. Γενικά ως ομάδα πάντως θα εγκρίνουμε τις τροπολογίες ε, πιθανότατα με την εξαίρεση κάποιων διατυπώσεων, για παράδειγμα εκεί που μιλάμε για την αποφυγή των μεταφορών τις έννοιες της αποφυγής των μεταφορών. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε διότι η Επιτροπή Μεταφορών δεν μπορεί να μιλά για την αποφυγή μεταφορών. Μπορούμε να θέλουμε να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι μεταφορές ως προς το κόστος και το όφελος, αλλά όχι να τις αποφύγουμε. Επίσης, δεν πιστεύω ότι η ε, Επιτροπή Βιομηχανίας θέλει να ε, εξαλείψει την βιομηχανία ή η Επιτροπή Υγείας ε, να ε, ξεχαστεί η υγεία. Ε, πάντως γενικά ο προϋπολογισμός αυτός εφαρμόζεται με νέο, νέα διαδικασία και πιστεύουμε ότι είναι πολύ λογικός για τους λόγους που είπαμε και η όλη διαδικασία έχει γίνει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ η κυρία Γένσιν για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις του εισηγητή. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει υποβάλει έναν ε, προϋπολογισμό ρεαλιστικό και επικεντρωμένο στα προβλήματα επιδιώκουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να υπερασπιστούμε και που πιστεύω ότι μπορούν να περάσουν από την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για την συνεργασία του. Αποσύρω τις τροπολογίες μου διότι αντικατοπτρίζονται απόλυτα στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι τα θέματα που επιδιώξαμε, τα δικαιώματα των επιβατών, ε, το, ε, η ενιαία διεπαφή ε, για, για το κλείσιμο εισιτηρίων στα ταξίδια, αυτό, όλα αυτά αντικατοπτρίζονται όπως και η χρήση του ITS. Επίσης επικροτώ το πιλωτικό πρόγραμμα για ε, μια ενιαία διαπαφή μεταφορών ε, και κλεισίματος εισιτηρίων. Έτσι θα μπορεί κανείς ε, να κλείσει τρένο σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης με την ίδια διαπαφή. Η δική μας ομάδα θα στηρίξει τη γραμμή που ακολουθεί ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ, η κυρία Ντυράν για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Ρικέ για την πολύ καλή συνεργασία. Δίκιο έχει όταν λέει ότι στη τωρινή οικονομική συγκυρία είναι σημαντικό ο τομέας των μεταφορών να χρηματοδοτηθεί επαρκώς. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτά τα νέα μέσα που έχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση συνολικά είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη. Εμείς ε, καταθέσαμε μερικές τροπολογίες ε, για να υποστηρίξουμε την αηφορία σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, για να υποστηρίξουμε ένα model shift μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέσο το οποίο θα είναι πολύ χρήσιμο και θα μας βοηθήσει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αηφόρα εικόνα για τις μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξει ότι δεν θα υποστηρίξω αυτά που έχουμε μπροστά μας ε, στο βαθμό που τα υποστηρίζουν οι άλλες πολιτικές ομάδες. Εξετάζοντας τις τροπολογίες που βλέπω, ε, εγώ νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει χάσει τα λογικά του. Σε χρόνο που κάθε κράτος μέλος πρέπει να κάνει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, έχουμε εδώ προτάσεις αύξησης ε, των ε, εσόδων του παρόντο από κάθε κράτος μέλος. Αυτό είναι τρελό. Ε, και ήλπιζα ότι η θέση αυτή θα περιοριζόταν στην Επιτροπή μας, αλλά από ό,τι φαίνεται ε, την ε, ακολουθεί όλο το Κοινοβούλιο. Και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου θα ήθελα να αυξηθούν οι δαπάνες. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα εδώ δεν είναι η αύξηση το, της χρηματοδότησης προγραμμάτων. Ε, οι περισσότερες αυξήσεις αφορούν αύξηση της γραφειοκρατίας. Ε, μιλάμε για αύξηση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών που έχουν δημιουργήσει. Και τι θα κάνουν όλα αυτά για τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ελάχιστα από ό,τι μπορώ να κρίνω εγώ και από, από ό,τι μας έχει δείξει η ιστορία. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία όπου μπορώ να θεωρήσω ότι ναι, δίνουμε χρήματα ε, σε κάπου που να αξίζει τον κόπο, αλλά η πλειοψηφία των αυξήσεων που βλέπουμε εδώ πέρα αφορούν αύξηση της γραφειοκρατίας και των γραφειοκρατών που ήδη υπάρχει. Η ομάδα μου λοιπόν δεν θα υποστηρίξει τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους και και τον εισηγητή φυσικά και να ζητήσω δύο διευκρινήσεις από τον εισηγητή. Βλέπω ότι 6406 τροπολογία όπου λέμε να προσέξουμε περισσότερο τα προβλήματα ασφάλειας των ποδηλατών στον δρόμο του Σαντιάγκο της Κομποστέλα, δηλαδή των ποδηλατών προσκυνητών εννοεί ο Μιλήτρια, Έχουμε λοιπόν εμείς αυτή την πρόταση και θέλουμε να την κρατήσουμε όπως ήταν και στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Θέλουμε λοιπόν να διατηρηθεί. Μετά, συμβιβασμός 1. Βλέπω ότι ο εισηγητής κάνει περικοπές στον κοινωνικό τουρισμό. Έχουμε αύξηση του τουρισμού 9% αλλά από την 1η Ιανουαρίου και μετά μετά δηλαδή τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι πλέον κοινή αρμοδιότητα ο τουρισμός θα ήταν πραγματικά ένα τραγικό πολιτικό μήνυμα να μειώσει αυτή η Επιτροπή τον κοινωνικό τουρισμό. Αν αρχίζουμε εμείς δηλαδή πραγματικά στην διαδικασία του προϋπολογισμού να περικόβουμε εμείς το ελάχιστο, ε, πραγματικά θα, θα, θα μια καταστροφή διότι όταν εμείς βάλουμε ένα ποσό ή ήδη βάζουμε ένα ποσό στην Επιτροπή μας και μετά πάει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ούτως ή άλλως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το κόβουνε άρα βάζουμε ένα εκατομμύριο θα μας το κόψουνε Ας το αφήσουμε λοιπόν όπως είναι, γιατί ούτως ή άλλως η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα μας το κόψει. Και ξέρουμε καλά ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και πέρα των καλών προθέσεων του Κοινοβουλίου που θέλει να κρατήσει τα ποσά, κόβονται μετά αυτά τα ποσά. Και ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα που ο Επίτροπος Σταγιάννη το έθεσε ως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και να βελτιώσει δηλαδή τη βιομηχανία του τουρισμού και τη βελτίωση των τουριστικών ροών στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε όλους τους ομιλητές στον κατάλογο. Μπορούμε λοιπόν να επανέλθουμε στον εισηγητή. Και να σας ε, θυμίσω ότι θα χρειαστείτε τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας σας για την ψηφοφορία. Όποιος λοιπόν δεν την έχει, έχει τώρα κάνα δύο λεπτά να πάει να τη, να, βρει. Ε, προτού να δώσω το λόγο όμως στη, στον Ντόμινικ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι που θέλει να πει. Euh, Συμφωνούμε με την έκθεση του κυρίου Ρίκε και δεν έχουμε άλλες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Δομινίκ. Ε. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους και οδησυγητές με τους οποίους εργαστήκαμε και ρεαλιστικά και ευχάριστα. Ήταν επικοδομητικότατη η συνεργασία τους. Ευχαριστώ λοιπόν. Δεν έχω πολλές παρατηρήσεις να κάνω. Ξέρετε όμως ότι είναι πάντοτε πολύ δύσκολη η δουλειά, ε, ο συνδυασμός μεταξύ των ε, ε, γενεόδωρων και των τσιγκούνιδων. Στις διοικητικές δαπάνες εμείς κοιτάξαμε να περικόψουμε τον προϋπολογισμό, δηλαδή προσέξαμε να μην διατηρήσουμε ε, μία γραφειοκρατία δαπανηρή και συντηρήσαμε τα λειτουργικά προγράμματα τον Κέσσαρα, τον Μαρκοπόλο που είναι προγράμματα πολύ λειτουργικά και αφο, δεν φύγουμε σε τίποτα το λειτουργικό στόχο των προγραμμάτων μας. Τώρα για τα υπόλοιπα συμφωνούμε. Τώρα για να απαντήσω στην Ινέσκα για το 6406. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Δεν θα την ε, κουτσουρέψουμε εμείς. Και ανέφερα εγώ τις ε, γενικές ε, θέσεις για τα προγράμματα, διατύπωσα εγώ μια θέση σχετικά μπορούμε να αυξήσουμε το κονδύλιο, μπορούμε να ψηφίσουμε σχετικά για τον συμβιβασμό 1 και για την 6406 δεν κατάλαβα εγώ αυτή την, εξυπορο... την εξισορρόπηση μεταξύ του 1, του 2 και του 08 δεν έχω άλλα σχόλια Μπορούμε να ψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Ντόμινικ. Να ευχαριστήσω όχι μόνο εσένα, το προσωπικό σου και τη γραμματεία και τους σκιώδεις συζητητές αλλά να ευχαριστήσω και τους βοηθούς τους για την σκληρή δουλειά που συνεπάγεται πάντα τέτοιου τύπου διαδικασία. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αυτή τη φορά διότι έχουμε μόνο μία ανάγνωση. Είμαι λοιπόν ευγνώμων για όλη τη δουλειά που έχει γίνει από εκλεγμένους και μη εκλεγμένους ε, ανθρώπους. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα θα κάνουμε μία δοκιμή. Όποιος ε, δεν έχει ε, κάρτα ή, δεν, ε, ή έχει χάσει ή τις έχει βάλει στο πλυντήριο ε, ή στο στεγνοτήριο. Σας παρακαλώ κατά τη διάρκεια της δοκιμής να μου το πείτε. Αρχίζουμε λοιπόν την δοκιμαστική ψηφοφορία. Όποιος δεν έχει την κάρτα του παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του να δούμε που βρίσκεται ο κύριος Αλκαντράουε. Ε, μας δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και ο Ντόμινικ, Έχουμε δύο ψήφους παραπάνω για το EFT. Παρακαλώ να το έχετε αυτό ε, κατά νου. Και όπως ε, είπα, παρακαλώ όσοι δεν έχετε κάρτες ε, να μου κάνετε νόημα με το χέρι όταν θα ψηφίζουμε. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 6406. 6406 υπέρ. κατά αποχές να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας λοιπόν για το, την τροπολογία 6406. ο κύριος Σαΐτ Αλκατράου και ο κύριος Ντομινίκ μου κάνουν νόημα. Έχουμε έναν πράσινο παραπάνω και δύο παραπάνω από το EFT. Το EFT που βρίσκεται. Δεν θα το κάνουμε αυτό μηχανικά λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι το μηχάνημα έχει κάποιο πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και πάλι. Ψηφίζουμε για το 6406. Ζήτω συγγνώμη το προσωπικό, θα πρέπει να μετρήσουν. Ποιο είναι υπέρ λοιπόν, σα παρακαλώ, σηκώστε ψηλά το χέρι σα. κατά. Απορρίπτεται. 6408 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6409 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6430 υπέρ. Κατά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 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 04 ματέρα ε, υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 05. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 και 31 αποσύρονται. 23. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, 26 ε, συγγνώμη, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 07 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογίες ε, του σχεδίου γνωμοδότησης. 1. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο είναι χωρισμένοι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το, όλο το κείμενο εκτός από τις έννοιες αποφυγής των μεταφορών. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος. Καταπίπτει. Τρίτη τροπολογία. Αγιάλα Σέντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. διράν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Σε δύο μέρη. Δεν είμαι βέβαιος πώς θα γίνει ο συμβασμό εφόσον είναι χωρισμένη. Το... Συμβαστική τροπολογία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το πρώτο μέρος είναι το ολόκληρο το κείμενο εκτός από την πρόταση που ενθαρρύνει τις μεταφορές με πολλά μέσα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος θα το ψηφίσουμε αυτό. Ναι, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Νόμιζα ότι η κυρία Γιάννησεν είχε αποσύρει όλες τις τροπολογίες της. Παράγραφος 6α, κυρία ε, Γιάννησεν, έχω εδώ ένα σημείο που λέει ότι θέλετε να κάνετε προφορική τροπολογία, σωστό? Από ό,τι γνωρίζω, λέει η κυρία Μάισνερ, η κυρία Γιάννησεν απέσυρε τις τροπολογίες που υπέβαλε μόνη τη. Αυτή εδώ όμω είναι μαζί με τον εισηγητή. Ρωτήστε λοιπόν τον Ντομινίκ. Από ό,τι φαίνεται είναι μέρος του συμβασμού. Ντομινίκ. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γένσεν για αυτή την προσθήκη. Το κείμενο βρίσκεται στο τέλος ε, του καταλόγου ψηφοφοριών. Θα το ψηφίσουμε αυτό λοιπόν μαζί με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει με την τροπολογία της κυρίας Σουεντιρό. Μιλάμε για διαφάνεια. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ωραία, φτάνουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Θα πρέπει να μετρήσουμε, παρακαλώ λοιπόν σηκώστε ψηλά τα χέρια σας, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πιο εύκολο αυτό. Κατά. Αποχές. Τριάντα μία ψήφοι υπέρ, τέσσερις κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Ρικέ για τη δουλειά σας. Να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας. Φαίνεται ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα με την ε, συσκευή για τις ψυχοφορίες. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση διερεύνησης συμβάντων και ατυχημάτων στην πολιτική αεροπορία. Προτού να δώσω το λόγο στη συγκύτρια κυρία Ντιβέρα. Θα ήθελα να θυμίσω στην Επιτροπή ότι η Διαπραγματευτική Επιτροπή ε, και σκιωδών εισηγητών έχει καταλήξει σε 93 ε, τροπολογίες που υιοθετήθηκαν και η κυρία Ριβέρα παρουσίασε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Στηρίξαμε τη δουλειά που έχει κάνει και τους συμβιβασμούς στους οποίους κατέληξε. Τώρα λοιπόν η κυρία Ριβέρα θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο σύνολο της Επιτροπής. Πρωτού λοιπόν σου δώσω το λόγο Κριστίν, θα ήθελα. Ευχαριστώ που κάνετε ησυχία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όσοι θέλετε να έχετε ιδιαίτερη ε, συζήτηση να τις κάνετε έξω από την αίθουσα. Υπάρχει πολλής χώρος. Ναι, για να ακούσουμε την κυρία Τιβέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου παρέχετε να έρθω εδώ και να συζητήσω σχετικά με την πρόοδο των εργασιών που έχουν εκπονηθεί ε, σε επίπεδο έρευνα ε, για την πρόληψη των ατυχημάτων στην αεροπορία. Μετά από αρκετέ εβδομάδε δύσκολων ε, διαπραγματεύσεων, πριν το καλοκαίρι φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να έχουμε μια πρώτη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την αποδοχή του αυτή τη συμβαστική πρόταση με επιστολή του τη 30η Ιουνίου ε, τρέχοντο έτου από τον πρόεδρο του Κορεπέ, τον Μπάρεν Σίμψον. Σύμφωνα με το άρθρο 70.3 του κανονισμού λειτουργία μα, σήμερα υποβάλλω υπόψη σα την συμβαστική αυτή πρόταση και ζητώ την στήριξή σα επί των αποτελεσμάτων ε, εάν ε, είμαι μεν ευχαριστημένη που βρήκα έναν τρόπο να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση, αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι το κείμενο που έχουμε σήμερα αναχείρας. Ε, είναι ένας κανός, είναι ένας καλός κανονισμός, απηχεί ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα έρευνας επί των ατυχημάτων και την ανάληψη των αποζημιώσεων για τις οικογένειες των θυμάτων. Ευχαριστώ τους σκιώδεις ε, εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που μας παρέσχουν ε, και που μας επέτρεψαν να καταλήξουν τα καλά τα αποτελέσματα. Σας ε, παρουσιάζω τις γενικές γραμμές της συμφωνίας και τις βασικές αλλαγές στο κείμενο αυτό, ε, ύστερα και από την υποβολή του Τραν περί τον περασμένο Ιουνίο. Ε, με την συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Εναέρης Κυκλοφορίας μπορέσαμε να διατηρήσουμε τον όρο του advisor πετύχαμε να πείσουμε το Συμβούλιο να άρει το στοιχείο της ανασφάλειας δικαίου που υφίστατο ε, στην γενικότερη προσέγγιση με τον όρο when relevant, όπου αυτό είναι πρόσφορο και εξάλλου ε, ένα εχέγγυο που διατηρεί τον κίνδυνο ε, για την σύγκρουση συμφερόντων που ε, παρέμεινε. Αυτή ήταν οι χειρονικέ γραμμέ, η σημαντική πρόταση που έγινε σε σχέση με την Επιτροπή. Όσον αυτό το επίπεδο εφαρμογή του κανονισμού, το Συμβούλιο θα ήθελε να τον συστάλλει. αυτό βέβαια θα σήμαινε μια υποχώρηση σε επίπεδο ασφάλεια ενέργεια κυκλοφορία. τελικά η άλλη θέση όμω κατήσχησε και η θέση τη Τραν επικυρώθηκε επί των ε, λόγων το Συμβούλιο επέμεινε σε κάποιες τροπολογίες ως προς την διοργάνωση του, του δικτύου χωρίς να επιβαρυνθεί το δίκτυο και να προσδοθεί ευελιξία. Δεν ήταν τα σημαντικότερα αυτά τα σημεία τροπολογίες, ωστόσο το σωστικό για τη δική μας Επιτροπή ήταν να προσδιοριστούν επακριβώς οι λειτουργίες του ε, δικτύου να θεσπιστούν οι αρχές ε, του ετησίου προγράμματος δράσης και να, να παρασχεθούν τα εχέγγυα για τη λειτουργία του κανονισμού. Τα τρία αυτά σημεία συγκερνώνται στο άρθρο 7 του κανονισμού. Όσον αφορά τις σχέσεις ε, της δικαστικής ερεύνας των τεχνικών ερευνών ασφάλειας, ένα θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο πολλών τροπολογιών σε επίπεδο τραν, ένα σημείο ιδιαίτερα ευαίσθητο για μας, προβλήματα σημαντικά ετέθησαν όσον αφορά την διαφορετικότητα των δικαστικών συστημάτων των 27 κρατών μελών. Στη συνέχεια η δυναμία επί της αρχής ε, ε, εξασφάλισης ε, πρόσβασης σε κάποια κείμενα χωρίς να προκειμένως να τροποποιηθεί το σύνταγμα κάποιων κρατών μελών. Να έχω κατά νου για παράδειγμα την Σουηδία που αυτό ισχύει και τέλος η αδυναμία σε πλαίσια ενός κανονισμού να υπάρξει νομική και πολιτική βάση για την τροποποίηση κανονισμών σε δικαστικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Για το λόγο αυτό, σε συμφωνία και με τον ε, Σκιώδη ε, εισηγητή, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στα δύο πρώτα σημεία. Μπορούμε εκεί να είμαστε αποτελεσματικοί, ήτι πρόσβαση των ε, ερευνητών ασφάλεια στα αποδεικτικά στοιχεία και ε, την σύναψη προσυμφωνιών μεταξύ των δικαστικών αρχών και των φορέων έρευνα. Όσον αφορά την πρόσβαση των ερευνητών στα αποδεικτικά στοιχεία, αποφασίστηκε ότι ακόμα και στα κράτη εκείνα όπου οι δικαστικέ αρχέ είναι εκείνε που έχουν τα αρμοδιότητα Μεταφορά και διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, ο τεχνικό Ερευνητή θα έχει και πάλι μια άμεση πρόσβαση ε, και απεριόριστη αποδεικτικά στοιχεία. Επί του προσυμφώνου που ήταν σημαντική τροπολογία που έγινε δεκτή σε επίπεδο τράνου, το κείμενο μα έγινε δεκτό και μάλιστα επιρώθηκε με προσθήκη τη υποχρεωτική ε, διαβίβαση των προσυμφωνών προ το Κοινοβούλιο, προ ενημέρωσή του. Ε, βρέθηκε λοιπόν συμβαστική λύση και είναι ικανοποιητική θα και από του σημείου αυτού. Όσον αφορά περαιτέρω το ζήτημα των ε, κατανάθεση πράξεων, ε, το Συμβούλιο ήταν πολύ επιφυλακτικό προ αυτό. Ήθελε να ε, υπάρξουν προποθέσει που θα προσέγγιζαν περαιτέρω αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη από ότι ένα, ένα άλλο όργανο με τον Σκιώδη. η συγητέ βασίσαμε ότι μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί ίσω ένα προηγούμενο για, για μελλοντική νομοθέτηση ενώ η κατανάθεση πράξη είναι η μόνη διαδικασία για δρομολόγηση νομοθετήσεις που δίνει ε, αρμοδιότητα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Προτάθηκε λοιπόν να αρθούν ε, μια και έξω όλα τα άρθρα περί των ε, κατανάθρωση πράξεων. Το Συμβούλιο τελικά το απεδέχθη αυτό. Με τον τρόπο αυτό παράσχουν τα εχέγγυα ότι σε περίπτωση τροπολογία του οργανισμού πρέπει να περάσουμε από την συναπόφαση και αυτό επιτρέπει στο δικό μα όργανο να έχει ισότιμη θέση με το Συμβούλιο. Επί του ζητήματος ε, της προθεσμία δημοσιεύσεω ε, ε, του καταλόγου επιβατών, η Επιτροπή μας και το Συμβούλιο ψήφισαν υπέρ της προθεσμίας των δύο ώρων. Η προθεσμία αυτή επικυρώθηκε, οπότε η υποχρέωση δημοσίευσης άμεσης του καταλόγου των επικινδύνων εμπορευμάτων παρόντων επί του ε, αεροσκάφους που υπέστη το ατύχημα προσθέθηκε. Όσον αφορά το αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων, πολλές τροπολογίες που έγιναν δεκτές στο Συμβούλιο δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό απέναντι στις τροπολογίες αυτές. Πάντως κάποιες ε, ελάσσον σημασίας τυπικής υφής τροπολογίες έγιναν δεκτές, ώστε όλα αυτά τα σημεία να απηχούνται στην συμβαστική πρόταση όπως για παράδειγμα στην, κατά τη φάση τη κράτηση θέσης να υπάρχει, ε, υπάρχουν τα στοιχεία για την ειδοποίηση σε περίπτωση ατυχήματο, η δυνατότητα προώθησης ε, εκ μέρου τη οικογένεια ε, ε, πληροφοριών σχετικά με την έρευνα πριν αυτό εμεσυρθούν. Εάν η οικογένεια το ζητήσει πληροφορίε για το άτομο επί του αεροσκάφου, ε, η υπόδειξη των ατόμων που ε, σε περίπτωση ατυχήματο θα παίξουν τον ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ του θύμα, της οικογένειας του θύματος και των αρμοδίων φορέων και αρχών σε περίπτωση έρευνας η υποχρέωση για όλες τις αεροπορικές εταιρείε ε, που έχουν εγκατάσταση στην Ευρώπη να διαθέτουν ειδικό ε, πλάνο κρίσης σε περίπτωση ατυχήματος ειδικά σε επίπεδο ψυχολογικής προστήριξης των οικογενειών των θυμάτων και τέλος η υποχρέωση όλων των εταιρεών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να έχουν μια ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων. Το τελευταίο σημείο της συμφωνίας έγκυται στο θέμα του απολογισμού των ε, περιστατικών cross-reporting ήταν το πιο δύσκολο από τα σημεία που είχαν διαπραγματεύσει. Ε, κάποια κράτη αντιτίθονται στην όλη αναφορά του στον κανονισμό αυτό. Με τον ε, ε, Σκιώδη εισηγητή ήμασταν πολύ στεναροί στο να υποστηρίξουμε το σημείο αυτό, γιατί ήταν η μόνη ευκαιρία να βελτιωθεί η πρόληψη των ατυχημάτων και ήταν αυτό απαραίτητο να υπάρξει αυτή η ευκαιρία ακριβώ για να υπάρχει δυνατότητα Πραγματική βελτίωσης του επίπεδου ε, ασφάλεια στην αέρα κυκλοφορία μετά από μακρέ διαπραγματεύσει, χάρη και στην υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο επεδέχθη την αρχή να παρέχονται προσβάσει στη βάση δεδομένων προκειμένου για τα ατυχήματα σε επίπεδο ΑΙΖΑ και στι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Επίση, έγινε δεκτό όπω αυτή η βάση δεδομένων τύχη ανάλυση προκειμένου να υπάρξουν προληπτικέ ενέργειε και να αποτρέπονται ατυχήματα στο μέλλον. Εξάλλου, ε, στην εντολική σκέψη που ο κ. Πρόεδρος ε, προέτεινε και που ζητούσε, ε, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει αναθεώρηση της οδηγίας ω προς τον απολογισμό των ατυχημάτων πριν την 31η Δεκεμβρίου 2011 και το σημείο αυτό έτυχε αποδοχή από το Συμβούλιο. Αυτό Αυτά ήταν εν πολύ στα κύρια σημεία της συμβατικής πρότασης. Να υπογραμμίσω ότι πραγματικά προσπαθήσαμε και δουλέψαμε σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασία με τον ε, και η προτινόμενη συμφωνία ε, σέβεται το πνεύμα που η Επιτροπή Τραν από 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους είχε κάνει δεκτό. Για το λόγο αυτό προτείνω να αποδεχθούμε, να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό και να το προωθήσουμε στην Ολομέλεια προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εξευρεθή σα συμβαστική λύση και ε, ήδη τη 4 Σεπτεμβρίου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στον Ομέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τιβέρα. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να πάει στην ε, Ολομέλεια της Δευτέρας, στη, δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ε, από τους χιλιάδες συγγητές, ε, από τους σοσιαλιστές και Σανκά. o Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη θέση μας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι παρατηρήσεις που έκανε η ομάδα μας έχουν ληφθεί υπόψη και πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλά ισορροπημένη η έκθεση αυτή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ από το, τους ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επανειλημμένα έχω ευχαριστήσει την εισηγήτρια στο όνομα της ομάδας μας. Είναι πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Θα ήθελα να την ξαναευχαριστήσω. Είναι κυρίως σημαντικό το ότι καταφέραμε μαζί με την Κομισιόν και ενάντια στο Συμβούλιο να επιμείνουμε ε, στην ε, περαιτέρω έρευνες, ε, στην πρόληψη των αεροπορικών ατυχημάτων στο μέλλον. Επίσης σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και να ε, προστατεύσουμε τους, ε, τους ε, επιβάτες. Ελπίζω να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό με ευρία συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρίχτεμπεργκερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ήταν πολύ θετική η συνεργασία που είχαμε. Τελικά, καταφέραμε κάποια θέματα που ε, μας ενδιαφέραν όλους ε, να τα περάσουμε. Δεν πίστευα ότι σε θέματα ασφαλείας παίζει τόσο σημαντικό ρόλο εγωισμός. Ε, ακούγοντας το Συμβούλιο, εξεπλάγην. Τα κράτη-μέλη πάντα πιστεύουν ότι αποκλειστικά και μόνο αυτά κατάφεραν να τετραγωνίσουν τον κύκλο και έχουν κάνει τρομερές ανακαλύψεις. Τελικά πάντως ε, ήταν καλός ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε, δεν ήταν εύκολο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών και το θέμα των ε, συγγενών των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος. Θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση για να συνοψίσω την κατάσταση. Αυτό που είδαμε εδώ ήταν η μεγάλη σύγκρουση σχετικά με ε, της πράξεις κατεξουσιοδότηση. Σε κάθε έκθεση θα αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, διότι το θέμα είναι εδώ ότι τα δικαιώματα ε, που έχει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε κάθε φορά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. διότι το Συμβούλιο προσπαθεί είτε από την πίσω πόρτα ε, προσπαθεί από την πίσω πόρτα είτε να αποδυναμώσει είτε να παρακάμψει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν ε, να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι το Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό και σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Και να είμαστε πιο πολύ με το μέρος των εμπειρογνωμόνων παρά με το μέρος των εθνικών λόμπις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα στο όνομα του ε, ECR να ευχαριστήσω την κυρία Ντεβιέρα για την ε, συμμετοχή των ε, σκιωδών εισηγητών και για τις συζητήσεις που είχαμε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι Ελπίζω για ε, μελλοντικές τεχνικές εκθέσεις σε θέματα όπως αυτό και δεν μιλάμε μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές ε, και για άλλες μορφές μεταφορών μιλώ. Θα ήθελα η σύνταξη να γίνεται με καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι η κυρία Ντεβιέρα είχε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει κατά την τροποποίηση του κειμένου αυτού και φαίνεται αυτό από τον αριθμό των τροπολογιών. Φυσικά υπάρχει η πολιτική διάσταση Κυρίως όμως επρόκειτο για τεχνική, τεχνικό κανονισμό. Ας ε, προχωρήσουμε λοιπόν από εδώ. Ε, παρακαλώ την Κομισιόν όμως να το σημειώσω αυτό. Άλλωστε έχουμε πει ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την, ε, τις αεροπορικές μεταφορές. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να είναι σωστά και σαφή τα κείμενα. Πάντως όπως είπε η κυρία Ντεβιέρα πολύ σωστά υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δείξαν σε συγκρούσεις, ε, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες νομικές και δικαστικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω πάντως ότι γενικά η, η διατύπωση στην οποία καταλήξαμε ήταν πολύ καλή. Επίσης ε, ήταν δύσκολο το θέμα σχετικά με την ε, υποβολή εκθέσεων. Ε, θα πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός. Ήταν πολύ σημαντικό και πολύ σωστό. ότι τελικά το Συμβούλιο άκουσε το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο άκουσε ε, και το Συμβούλιο, διότι όσοι ασχολούνται με τα θέματα των ε, αεροπορικών ατυχημάτων ε, έχουν συνεργαστεί πολύ στενά και με τους Υπουργούς και με την Επιτροπή μας για να βεβαιωθούν ότι θα έχουν καλό αποτέλεσμα με την έκθεση αυτή και να μην πρέπει να επανέλθουν στην Επιτροπή μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γενικά λοιπόν ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό. Έχουμε πολύ καλές ε, διαδικασίες ασφαλείας ε, στα κράτη-μέλη. Έχουμε πολύ καλές ομάδες ε, διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων και νομίζω ότι μπορούμε να επωφεληθούμε όλοι. Επίσης όσον αφορά την ενημέρωση των επιβατών που ανέφερε η κυρία Τεβιέρα, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να επικροτήσουμε ότι έχει συμπεριληφθεί με πολύ καλό τρόπο στην έκθεση και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει καλά στην πράξη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και θα στηρίξει η ομάδα μας την έκθεση αυτή στην δεύτερη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω και εγώ την, για την καταπληκτική αυτή εργασία που έχει γίνει στο φάκελο αυτό. Πολύ απλά θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσει και μετά να σε ένα σχόλιο. Πρώτο ερώτημα αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ενεργή Ασφάλεια όπως κατάλαβα, όπως προτάθηκε, ακριβώς διατηρείται η προτινόμενη αυτή υγειονομική φύσεως ε, διαχώρηση μεταξύ της έρευνας και της πιστοποίησης. Θα ήθελα να ξέρω, εάν έχει ε, προβλεφθεί, θα υπάρξει ένα feedback σχετικά με την τεχνογνωσία. Ε, με αφιτηρία ακριβώ τι έρευνε αυτέ ε, υπάρχει κάτι τέτοιο, για μένα είναι απαραίτητο και έχει μεγάλη σημασία ώστε και η ΕΣΑ να μπορέσει να το αξιοποιήσει στα πλαίσια τη διαδικασία πιστοποίηση και τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών. Έχει προβληθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, οι ερευνητέ. Μιλάμε πάντα για εθνικέ αρχέ. Γνωρίζετε πολύ καλά, ωστόσο, ε, ύστερα και από τα πρόσφατα ατυχήματα των αεροπορικών εταιριών στην Ισπανία, παρεμβαίνουν και αρχές που δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. Ε, μιλάμε για ερευνητικού φορείς από την πλευρά των εταιριών, οι δήμονες, Ευρωπαίοι κτλ. Θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο διερευνάται η εμπλοκή και αυτών των φορέων και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο δραστηριοποίηση αυτών των ερευνητών που εντάσσονται στην ερευνητική διαδικασία και που συχνά βλέπουμε να έχουν προβλήματα ε, και συνεργασίας. Επίσης, ε, τι θα γίνει σχετικά με την προστασία των εμπλεκομένων αυτών ατόμων σε ένα ε, όχι όμως επιβατών, όπως είναι τα πρόσωπα που δουλεύουν στη συντήρηση των κυβερνητών. Πώς θα υπάρξει προστασία αποτελεσματική και των κατηγοριών αυτών. Μιλάμε για την πρόληψη βέβαια σε επίπεδο αξιοποίησης αυτών των στοιχείων με ζωτική σημασία θα γίνει αυτό με τρόπο ώστε τελικά να αποτραπούν οι κίνδυνοι. Δεν μιλάω βέβαια για παράνομες ενέργειες, γιατί προφανώς μια τέτοια διαδικασία περνά άμεσα από τις δικαστικές αρχές. Αλλά με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία προστατεύουμε και εμείς τα άτομα αυτά που με τη σειρά τους παρέχουν τα για μεγαλύτερη ασφάλεια στην νέα κυκλοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκπρόσωπό τη να ε, λάβουν το βήμα, θα ήθελα και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή ε, προσπάθεια, το αποτέλεσμα τη εργασία τη και την αγαστή συνεργασία που είχε με τον εισηγητή και με ένα προσωπικά για το συντονισμό αυτή τη προσπάθεια, για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και για όλα αυτά. Επίση, να πω ότι θα ήθελα να ακούσω και άλλε απόψει, ακόμα και αν δεν συγκεραστούν, ακόμα και αν δεν ληφθούν υπόψη, είναι γόνιμο να λάβουμε υπόψη μα όλε αυτέ τι προτάσει Οτιδήποτε προτείνεται προ τον Σκιώδη εισηγητή και του υπολείπου έχει αξία. Προσωπικά λοιπόν θα ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την μακρά και επίπονη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού είναι Κύριε παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημερίζω όλους και όλες. Θεωρώ ότι και από τις παρεμβάσεις και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από την εισηγήτρια αλλά και από τον σκιώδη εισηγητή σήμερα το πρωί μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο ιδιαίτερα δύσκολος αυτός τομέας πλησιάζει πλέον σε μια πρώτη επιτυχία μέσω της πρώτης ανάγνωσης και ίσως μια λύση. Από την πλευρά της Επιτροπής εμείς εγκύπτουμε στις αρχικές θέσεις ε, του Ευρωκοινοβουλίου, της ε, Επιτροπής και του, Συμβουλ, του Επιτρόπου ε, επί των θεματών της, των μεταφορών. Συνυπογράφω λοιπόν τα συγχαρητήρια προς τον εισηγητή και, την, και τον ισχυρό εισηγητή για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν. Καθ' τουλάχιστον αυτό διασφαλίζει την προστιθάμενη αξία που από την αρχή επιζητούσαμε να υπάρξει ήδη κατά τη συντακτική φάση αυτής της πρότασης. Ουσιαστικά έχουμε καλύψει ό,τι έπρεπε να καλύψουμε και για να είμαι πιο σωστός για διατύπωσή μου μας ενδιαφέρει ένα σύστημα που να προσλάβει μια σαφή ευρωπαϊκή ε, διάσταση όσον αφορά την έρευνα, όσον αφορά ε, το σύστημα που θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο δραστήριοι σε επίπεδο πρόληψης ε, των ε, ε, αεροπορικών στο μέλλον. Κάτι που άλλωστε και ο συγητής υπογράμμισε, αλλά και εγώ θα το τονίσω, πρέπει καταρχήν, και να σας το πω, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προλαμβάνοντας μια πρώτη συμφωνία αργότερα μέσα στο μήνα, ήδη έχει δρομολογήσει την τεχνική προσπάθεια και τα όσα μένουν ακόμα να γίνουν στον τομέα αυτό. Προχωράμε λοιπόν, Προσβλέπουμε με ενδιαφέρον λοιπόν κύριε Πρόεδρε στην επιτυχία ε, και τη ψηφοφορίας κατά την δεύτερη ε, ολομέρεια του Σεπτεμβρίου και αν ε, μπορώ να συμπεράνω από την σημερινή μας συζήτηση υπάρχει ήδη ευρύτατη συνένεση από πλευρά των μελών της Επιτροπής ε, τα κράτη-μέλη έχουν τις συγκεκριμένες θέσεις και πολλοί θα το δεχτούμε. Δεν ήταν δύσκολο να υπερκεραστούν κάποιες πρώτε επιφυλάξει που αρχικά είχαν εντυπωθεί Συγχαίρομαι στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιτυχίες του διαπραγματεύσει. κάτι που μας φέρνει πιο κοντά στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα έτσι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εργασία αυτή. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ την κυρία Κριστίν. Ευχαριστώ. Ήδη το ρωτήσατε αυτό για τους πιλότους ΙΝΕΣ και σας είχα πει ότι θα υπάρχει μια απόλυτη μυστικότητα για τα στοιχεία που θα δώσουν οι πιλότοι στις έρευνες. Για τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφαλείας θα έχουμε μία τράπεζα δεδομένων που φυσικά θα αναλυθεί και θα χρησιμεύσει για να ληφθούν ε, προληπτικές δράσεις, για να μην έχουμε δυστυχήματα. Και φυσικά θα αναλύουν οι αρμόδιες αρχές ταυτόχρονα με την Άιζα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν συμφωνούμε λοιπόν όλοι, θα προχωρήσουμε με την υποβολή της έκθεσης ε, στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου τη δεύτερη. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εργασία της. Προχωράμε τώρα στις διάφορα άλλα θέματα. Δεν έχω κάποιες προτάσεις. Αν έχετε κάποια πρόταση τώρα μπορείτε να την υποβάλλετε για να τεθεί στα διάφορα άλλα θέματα. Εάν όχι, απλά να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη μας συνάντηση είναι Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ώρα 15 και 30, απαγευματινή Ζητώ από τους συντονιστές να είναι πίσω στις 10.30 και θα προχωρήσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών. Δεν μπορώ να ξεκινήσω νωρίτερα γιατί υπάρχει ε, προγραμματισμός. 10.30 ε, λοιπόν ξεκινάμε. Ευχαριστώ όλους και πάλι ευχαριστώ.